Ladies and gentlemen, can I, before we just start the meeting... Να αρχίσουμε τη συνεδρίαση. Να σας ενημερώσω ότι σήμερα είναι τα γενέθλια του κυρίου Ρικέ. Χρόνια πολλά κύριε Ρικέ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα τυπικά καταρχήν. Έχουμε ένα ξεχωριστό σχέδιο ημερήσιος διάταξης. Είναι κοινή συνεδρίαση της ΙΤΡΕ και της Transport. Τώρα συνεδριάζει μάλλον στο πλαίσιο της Επιτροπής Μεταφορών, συμφωνείτε επίσημα με τη Μέσια Διάταξη. Εισαγωγικά, να σας υπενθυμίσω ότι η έκθεση για την, το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη, τη διευκόλυνση μέσο για την Ευρώπη, θα παρουσιαστεί από τρεις εισηγητές με βάση το άρθρο 51 του καταστατικού του Κοινοβουλίου. Έχουν ένα σχέδιο έκθεση συντάξει και τρεις αυτοί συνεισηγητές. Είναι η σειρά της Επιτροπής Μεταφορών να φιλοξενήσει αυτή την κοινή συνεδρίαση. Την επόμενη φορά, όταν σκεφτούμε τις τροπολογίες της 5 Νοεμβρίου, η κυρία Σαρτόρη θα μας φιλοξενήσει σε αυτή την κοινή συνεδρίαση για τις τροπολογίες. Πριν δώσω το λόγο στους εισηγητές, θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Σαρτόρη μήπως έχει να προσθέσει κάτι, κάτι καινούριο. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη δουλειά που γίνεται και για τη δυνατότητα που μας δώσετε ε, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η πολιτική στιγμή ε, για την κοινή μας δουλειά. Έχουμε τρεις ε, εισηγητές από τρεις διαφορετικές χώρες, από τρεις διαφορετικές πολιτικές ομάδες που διαπραγματεύονται, που συζητάνε ένα τόσο σημαντικό θέμα στην δύσκολη αυτή πολιτική συγκυρία. Συγχαρητήρια για αυτούς τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν και σας περιμένω στην επόμενη συνεδρίαση. Αφήνω όμως τον πρόεδρο Σίμψον να ξαναπάρει τα ενία. Λοιπόν, σαν καλοί οικοδεσπότες, θα δώσω το λόγο στην κυρία Βαλιάν και συνεχεία στους άλλους δύο ε, εισηγητές. Παρουσιάζουμε από κοινού την έκθεσή μας σήμερα, μαζί με τους δύο συνεισηγητές. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για τη θαυμάσια συνεργασία τους τελευταίους εννέα μήνες και οι τρεις μας θα σας δείξουμε ότι το άρθρο 51 μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά. Ως εισηγητής, εισηγήτρια της ΣΥΤΡΕ θα σας μιλήσω για τη χρηματοδότηση του τομέα των τηλεπικοινωνιών και κοινωνιών και ενέργειας. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε πρωτοβουλίες υπέρ της ανάπτυξης, ούτως ώστε να αναζωογονήσουμε την οικονομία μας και τις ε, πολιτικές απασχόλησης και Καλωσορίζω λοιπόν το μέσο αυτό, τη διευκόλυνση αυτή. Η γενική φιλοσοφία, ε, συντάσσοντας αυτή την έκθεση, ήταν να πετύχουμε αυτούς τους στόχους με το πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ε, έχουμε λίγους πόρους στη διάθεσή μας, να χρησιμοποιήσουμε το καλύτερο τρόπο, να δούμε ποιες είναι οι κατάλληλες προτεραιότητες, οι πιο έκτακτες ανάγκες για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών υποδομών. Η ευρωπαϊκή πολιτική υποστήριξης ε, εξασφαλίστηκε στον τομέα ε, των μεταφορών μέσω της πολιτικής ευρωπαϊκών δικτύων. Και τα ευρωπαϊκά προγράμματα ε, χρηματοδοτούνται παραδοσιακά με δημόσια κονδύλια. Όμως, στον τομέα της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, πρώτη φορά τέτοια, μια τέτοια συγκεντρωτική στρατηγική προωθήθηκε και για να εντοπίσουμε προγράμματα με ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και για να επιτρέψουμε ε, σημαντική δημόσια χρηματοδότηση. Γι' αυτό θα πρέπει να δράσουμε πολύ προσεκτικά και υπεύθυνα, ιδίω σε αυτούς τους δύο τομεί, ούτω ώστε να αποφύγουμε ε, στρεβλώσει τη αγορά και να εξασφαλίσουμε την μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση των ελάχιστων πόρων που έχουμε ε, μέσω της επεκταμένης χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων. Έχουμε επενδυτικές ανάγκες που φτάνουν στα 1-3 ευρώ, 3 εκατομμύρια ευρώ για την ενέργεια, αν θέλουμε να εξυγχρονίσουμε και να επεκτείνουμε τις ευρωπαϊκές υποδομές. Η Κομισιόν υπολόγισε ότι 2000, ε, ε, μέχρι το 2020 δεν θα έχουμε τα κονδύλια που θέλουμε ούτε από το δημόσιο ούτε από τον ιδιωτικό τομέα για την ενέργεια και τις α, τηλεπικοινωνίες και τα 20 δισεκατομμύρια που δίνει αυτό αυτή η διευκόλυνση ε, καλύπτουν αυτό το επενδυτικό κενό χρησιμοποιώντας το πολυπλασιαστικό μοχλό ε, που προβλέπει αυτό το μέσο. Με, τις λίγες, ε, με το λίγο σπόρους χρειαζόμαστε ισχυρά μέσα μόχλευσης ούτως ώστε να κινητοποιήσουμε και ιδιωτικά κονδύλια. Δεν μπορούμε δηλαδή να βασιστούμε μόνο στις ε, δημόσιες επιχορηγήσεις. Γι' αυτό το μέσο της ενέργειας λέει ότι το 80% του προπολογισμού του μέσου θα πρέπει να δοθεί σε προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος μέσω χρηματοπιστωτικών μέτρων. Αυτά τα προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος θα πρέπει να είναι εμπορικά βιώσιμα, αλλά μπορεί να μην εξασφαλίσουν ιδιωτικού πόρους, γιατί ε, δεν είναι ελκυστικά πιστοτικά πώς. Φυσικά ε, θα χρειαστούμε κάποια επιδότηση, επιχορηγήσεις ε, για να κινήσουν αυτά τα προγράμματα. Θα πρέπει να εντάσσονται στην αγορά, να υπάρχει ασφάλεια των εφοδιασμού και ανανέωση των δικτύων ε, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, θα πρέπει να ζητήσουμε στις τηλεπικοινωνίες αύξηση της ζήτησης των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Γι' αυτό ε, θα πρέπει οι ψηφιακές υπηρεσίες της Ευρώπης να χρηματοδοτούνται, να έχουμε τις ακατάλληλες πλατφόρμες, οριζόντιες προτεραιότητες και την Ευρωπαϊκή μέσω επιχορηγήσεων. Επίσης, ε, οι ευρυζωνικές υπηρεσίες ε, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται με χρηματοπιστωτικό μέσα, προκειμένου να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση. Επίσης, θα πρέπει η αγορά να παραμείνει στο κέντρο της διαδικασίας για να μην έχουμε στρεβλώσει και για να αντισταθμίσει την, τον πολιτικό παρεμβατισμό. Το πιο δύσκολο καθήκον τώρα για μας είναι να πείσουμε το Συμβούλιο να εξασφαλίσει τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ που ανακοινώθηκαν ε, στις διαπραγματεύσεις ε, για τη διευκόλυνση, στο, στο μάλλον δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, τώρα όλα τα κράτη θέλουν να μειώσουν τον προπολογισμό και ειδικά τον προπολογισμό τέτοιων μέσων όπως το, η διευκόλυνση για την Ευρώπη. Αποφασίστηκε επίσης ε, να μην υιοθετηθεί η έκθεση συναπόφασης πριν να συμφωνήσουμε Πρέπει να ασκήσουμε όσο να περισσότερη πίεση σε αυτέ τι διαπραγματεύσει. Μην ξεχνάμε όμω ότι μπορεί να συρρυκνωθεί ουσιαστικά ο προπολογισμό. Πιστεύω ότι τι επόμενε εβδομάδε έχει γίνει μια σημαντική συζήτηση για να αποφασίσουμε ποια, ποιες είναι οι πιο ε, σημαντικές ε, προτεραιότητες στην ενέργεια και στις επικοινωνίες. Θα πρέπει να πολεμήσουμε και για τον προϋπολογισμό ε, της διευκόλυνσης, θα πρέπει, να επανεστιάσουμε τις προτεραιότητες με βάση τα μέσα. Αν τα μειωθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι, θα πρέπει να κάνουμε πιο δραστικές πολιτικές επιλογές, να δούμε τι θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε και τι να αφήσουμε στην πάντα. Στον τομέα της ενέργειας μπορεί να χρειαστεί να δώσουμε προτεραιότητα σε μία από τις τρεις διαστάσεις. Ε, ολοκλήρωση αγοράς, ε, ασφάλεια του ανεφοδιασμού ή ανανέωση των δικτύων ε, μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ε, επίσης, θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε ευρυζωνικά δίκτυα ή όχι. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Επίσης, ε, έχουμε και άλλους τομεί τομείς Θα πρέπει να βοηθήσουμε την ε, Κομισιόν να προσανατολιστεί στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Ε, είναι δύσκολο να επιλέξουμε, αλλά είναι ευθύνη μας να θέσουμε πολιτικές προτεραιότητες και να κάνουμε την πιο αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων. Περιμένω να γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ευχαριστώ και τους συνεισηγητές για τη θαυμάσια συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βαλεάν. Έρχομαι στου συνεισηγητέ από την Επιτροπή Μεταφορών. Θα αρχίσω από τον κύριο Ρικέ, όχι για κανένα λόγο, επειδή είναι τα γενέθλιά του. Και μετά, κυρία Γιάλα. Παρακαλώ, κύριο Ρικέ. Euh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους συνεισηγητέ. Δύσκολο βέβαια να είναι κανεί μόνο του με δύο ισχυρέ γυναίκε, αλλά Θα ήθελα επίσης να ε, ε, ευχαριστήσω τους σκιώδεις ε, εισηγητές και τους εκπροσώπους της Επιτροπής με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις που μου φαίνονται σημαντικές. Πρώτον, είναι ότι υποστηρίζουμε πλήρως αυτή την απόφαση της Επιτροπής. Δεν ε, είναι η πρόθεσή μας ε, στην, μέσω της έκθεσης να τροποποιήσουμε σημαντικά την απόφαση αυτή και θα ήθελα να το υπογραμμίσω. Κάποιες άλλες παρατηρήσεις. Πρώτον, η διευκόλυνση αυτή συνδέοντας την Ευρώπη είναι ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ανάπτυξη στην ε, Ευρώπη τόσο όσον αφορά την εργασία αλλά και την ε, δημιουργία υποδομών. Γιατί μέσω αυτών των υποδομών δημιουργούνται θέσεις εργασίας ε, και για τη δημιουργία αυτών των υποδομών και μετά στη βιομηχανία και μετά γενικότερα στην ενιαία αγορά. Αυτά είναι επίσης ε, υποδομές οι οποίες βοηθούν την ε, διασύνδεση της Ευρώπης και της ενέας ε, αγοράς συνολικά σε όλους τους τομείς, σε όλες τις ροές της ενέργειας των τηλεπικοινωνιών και συμβάλλουν στην ενοποίηση της ενιαίας αγοράς. Επίσης, μιλάμε τώρα για ένα, μια χρηματοδοτική διευκόλυνση. Και επιμένω σε αυτό, θα ήθελα να ζητήσω και από όλους τους συναδέλφου να το, ε, να το, έχουν υπόψη τους ότι θα πρέπει να είναι αυτό το, αυτός ο μηχανισμός ε, αποτελεσματικός Γι' αυτό θα πρέπει το κείμενο να παραμείνει ε, ε σαφές και συνεκτικό. Τα 50 δισεκατομμύρια που είναι το, τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας συνολικά. Πρέπει να κατανεμηθούν και η θέση του Κοινοβουλίου είναι ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε καταλήξει στη συνολική διαπραγμάτευση τίποτα δεν έχει κρυθεί. Δεν ε, θεωρώ ότι αυτό θα έχει νομοθετική επίπτωση στο δικό μας κείμενο, στο κείμενο που εξετάζουμε. η τελευταία γενική παρατήρηση. Συμφωνήσαμε με την κυρία Άγιαλα να μην ε, αγγίξουμε το θεζήτημα του παραρτήματος 1 στην έκθεσή μας και θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι θα παραμείνουμε, ε, θα εξετάζουμε το κύριο δίκτυο, το δίκτυο των κυρίων διαδρόμων και τα κριτήρια που είχαν συμφωνηθεί ε, θα πρέπει να εφαρμοστούν. Ε, παρά την ε, ίσως διάθεση που μπορεί να έχει κάποιος να προωθήσει περιφερειακά και σε ανησυχίες στο επίπεδο το ευρωπαϊκό. Τώρα στο ζήτημα της ενέργειας και των τηλεκοινωνιών. Θα θέλαμε να ενισχύσουμε την συνεκτικότητα αυτού του κανονισμού με την στρατηγική Ευρώπη 2020. Δηλαδή την ανάπτυξη, την ΕΦΗ, e, την αιφόρο και πώς θα γίνει αυτό. Να δημιουργηθούν ΕΦΗ e συστήματα μεταφορών, να αξιοποιηθούν τα ε, πολύτροπα συστήματα μεταφορών και την επιστροφή σε μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ισορροπημένη ανάπτυξη. Συμπεριλαμβάνοντας και τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Τώρα, σε συνδυασμό με τη στρατηγική 2020, Ευρώπη 2020, θα πρέπει να βρεθεί το σωστό επίπεδο συγχρηματοδότησης ε, των προγραμμάτων έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα διασυνοριακά δίκτυα που είναι απαραίτητα για την διασύνδεση των διαφορετικών περιοχών της Ευρώπης. Πρέπει να υποστηρίξουμε την πραγματική ε, ε, ενοποίηση και ολοκλήρωση των ε, κρατών εκείνων της Ανατολικής Ευρώπης που έχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα στο ζήτημα της συγχρηματοδότησης προγραμμάτων. Και αυτό το τμήμα της Ευρώπης πρέπει πλήρως να, να ολοκληρωθεί, να ενοποιηθεί με την υπόλοιπη Ευρώπη και αργότερα και με τις τρίτες χώρες, δηλαδή με τις χώρες οι οποίες βρίσκονται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό ε, ρυθμίζεται από, αυτό το από αυτή τη χρηματοδοτική διευκόλυνση, αλλά επίσης είναι σημαντικό τα ίδια τα κράτη-μέλη ε, ε, να βρουν εκείνο το στοιχείο που θα τα βοηθήσει να υλοποιήσουν τα δικά τους προγράμματα. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που έχουμε μείνει στο ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών και έχουμε επίσης επιμείνει στη σημασία της ενίσχυσης των συνεργειών μεταξύ αυτών των τριών τομέων της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σημαντικοί δημοσιονομικοί περιορισμοί για τους λόγους που σας εξήγησα το γεγονό ότι βρισκόμαστε στη, διάθεση, στη διάρκεια μιας ε, περίοδου, ας το πούμε, λιτότητας που ζητείται η εξορρόπηση των δημόσιων προπολογισμών αυτό θα... Ε, βρισκόμαστε μέσα σε αυτές τις συνθήκες και ακόμα ένας λόγος είναι αυτός για να έχουμε στη διαθεσή μας μια χρηματοδοτική διευκόλυνση, ένα μηχανισμό σωστά στημένο που θα βρει το, τη θέση του στο πλαίσιο πολιτικών που ήδη υπήρχαν και ήδη εφαρμόζονταν στο ευρωπαϊκό επίπεδο και που ήδη είχαν αντίκτυπο σε μεγάλο βαθμό στους προπολογισμούς και στην ε, ανάπτυξη και στην προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και από απ τα σημαντικά στοιχεία που υπογραμμίζουμε στη, στην έκθεσή μας, ο τρόπος με τον οποίο θα ενισχύεται η προστιθέμενη αξία κατά την επιλογή των προγραμμάτων. είναι πιθανόν να χρειαστεί περισσότερες χρηματοδότησης, περισσότερες επιδοτήσεις για ε, τις μεταφορές, γιατί συχνά δεν είναι, ε, μπαρκούν οι πόροι, αλλά επίσης θα πρέπει να αξιοποιηθεί η μόχλευση. Ε, ίσως αυτός να είναι ένας τρόπος να λύσουμε μια σειρά προβλημάτων. Να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε αυτούς τους δύο τρόπους χρηματοδότησης και την επιχορήγηση και να τις συμπληρώσουμε κατά μία έννοια με τα χρηματοδοτικά μέσα. Και όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, πρέπει να έχουμε ε, υλοποίηση των προγραμμάτων έτσι ώστε να λειτουργούν μέσα στην ε, χρονική προθεσμία που είχε τεθεί εξ αρχής. Ζητάμε πολλά, όπως βλέπετε, είμαστε πολύ φιλόδοξοι και ευελπιστούμε, αλλά για, αυτό το κάνουμε γιατί θεωρούμε ότι αυτό το χρηματοδοτικό μέσο είναι εξαιρετικά μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γιάλα Σέντερ. Τρίτη συνεισηγήτρια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τον κατάλογο μιλητών. Έτσι και μία ώρα έχουμε μόνο. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία ε, και τους δύο συνσηγητές συναδέλφους αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βοήθειά της. Είμαστε σε μόνιμη συζήτηση βεβαίως και τη γραμματεία μας αλλά και τον κύριο Σαγκάρ, ε, εισηγητή της Επιτροπής Περιφερειών, που είχαμε επανειλημμένες συναντήσεις μαζί του και τους σκιώδεις εισηγητές που ε, είχαν την καλοσύνη να μας δώσουν ε, μια πρώτη εντύπωση για την πρώτη μας πρόταση. Αυτή η άσκηση είναι ουσιαστικά πολιτική ε, δεδομένου του δημοσιονομικού πλαισίου και της συζήτηση με το Συμβούλιο. Και τώρα είναι η ώρα να κάνει αυτό το βήμα το Κοινοβούλιο υπέρ της επένδυσης, της ανάπτυξης, της μεγένθησης της οικονομίας, της απασχόλησης και της περισσότερης Ευρώπης, όπως πολύ ωραία είπατε. Αλλά και το ιστορικό είναι μια μεγάλη απογοήτευση, ματέωση ε, της Επιτροπής μας εδώ των μεταφορών. Κάθε φορά που προσπαθούσαμε να στήσουμε ένα σύστημα ε, επικοινωνιών με διευρωπαϊκά δίκτυα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με φιλοδοξία και ευρωπαϊκή και διασυνοριακή ε, προσκρούμε σε βίες περικοπές του Συμβουλίου. Δηλαδή αυτή η συζήτηση με το Συμβούλιο μας οδήγησε στο να κάνουμε μια άσκηση αρκετά περιοριστική στα ουσιαστικά όμως να δώσουμε ένα μήνυμα ότι αν δεν υπάρχουν περισσότερα χρήματα. Προς το παρόν θα περιοριστούμε στους διαδρόμους που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παράρτημα 1. Δηλαδή δεν θα πάμε παραπέρα με κάποιες εξαιρέσεις που ακούσαμε να διευρεθεί το θέμα των αστικών κόμβων και της πρόσβασης και επίσης ε, οι συνέργειες μεταξύ τουλάχιστον δύο από τους τρεις ε, τομείς που επεξεργαζόμαστε από κοινού και νομίζω αυτό θα είναι καλή ε, προσπάθεια για το μέλλον. Και να ανοίξουμε την πόρτα έστω και προσεκτικά στα νέα χρηματοδοτικά μέσα για τις μεταφορές, αν μη τι άλλο. Γιατί αν δεν αρκούν τα χρήματα, η Επιτροπή Μεταφορών θα προσπαθήσει ακριβώς να περιορίσει του προσπάθειες. Εξού και η ιδέα στην πρώτη πρόταση να μην θίξουμε τον κατάλογο που μας είχε δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχικά για να πούμε ότι αν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για περισσότερες ευρωπαϊκές υποδομές, έτσι, ευφυής όμως με άλλη φιλοσοφία, με άλλο σχήμα που να ε, είναι πιο αποτελεσματικό και πιο αξιόπιστο στα μάτια των πολιτών. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι πόροι θα περιοριστούμε στα ελάχιστα που ζητούμε. Θα υπάρξει μεγάλη πρόταση από ό,τι φαντάζομαι έτσι πλήθος προτάσεων των συνάδελφων. Προφανώς έχουμε ξεχάσει κάποια πράγματα ε, στα παραρτήματα. Έχουμε ήδη δει προτάσεις των συναδέλφων, αλλά εμεί θέλουμε να περιοριστούμε στη μεθοδολογία με τις κατευθυντήριες γραμμές που είπα και οι συνάδελφοι. Είναι καλή αυτή η μεθοδολογία με κάποια μικρή ίσως διόρθωση. Πάντως χρειάζεται επαρκής προϋπολογισμός για να καλύψει αυτές τις ανάγκες και να προωθήσει αυτό το θέμα. Και τελευταία, το Κοινοβούλιο συζητάει με το Συμβούλιο για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και θα θέλαμε να ε, εξαντλήσουμε τα όρια. Το είπαμε και με τον κύριο Ρικέ. Δηλαδή, αν δεν έχουμε χρήματα, να περιοριστούμε στη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η γελιότητα που ισχύει μέχρι τώρα. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε ακραίοι, γεριζοσπαστικοί στην προσέγγιση μας. Λοιπόν, ας μη σας εκπλήξει που είμαστε έτσι περιορισμένοι στις προτάσεις μας, γιατί θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα και πολιτικό μήνυμα. Ότι αν υπάρχουν πόροι, φιδωλά να τους ε, απορροφήσουμε, θα δούμε τις προτάσεις των συναδέλφων και Στι χώρε συνοχή, Κοιτάξτε τι τροπολογίε 27 και 72 και πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να είναι μια βάση για να οικοδομήσουμε μαζί με άλλες τροπολογίες της Περιφερειακής Επιτροπής που ήδη έχουν κατατεθεί για να δούμε αν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια φόρμουλα για να βελτιώσουμε και τα διευρωπαϊκά δίκτυα σε όλη την Ευρώπη και στις χώρες συνοχής. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον κύριο Πίπερ, που είναι της Περιφερειακής Επιτροπής Κιώδης, συντάκτης μάλλον, και μετά ο κύριος Ζάγκα από την Επιτροπή των Περιφερειών. Τρία λεπτά έκαστο, σα παρακαλώ κύριοι, αλλιώ δεν θα προκάνουμε. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα συζητάμε και οι διερμηνείς θα αποχωρήσουν. Ο ε, κύριος Πίπερ από την Περιφερειακή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την ουσία της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη, δεν θα μπω εγώ, επανειλημμένα τα ακούσαμε. Θέλω να σας επισημάνω το εξής. Η Περιφερειακή Επιτροπή έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τα χρήματα των Ταμείων Συνοχής και τα 10 δισεκατομμύρια που προβλέπονται μέσω των Ταμείων αυτών, του Ταμείου Συνοχής. Εμείς κάναμε λοιπόν το εξή βήμα ήδη. Όταν ψηφίσαμε το Γενικό Κανονισμό για τα διορθωτικά ταμεία, σε μια συμβιβαστική πρόταση, δυστυχώς η διαδικασία διαγωνισμών για τη συνδέοντα στην Ευρώπη αμφισβητήθηκε. Τα λέω πολύ προσεκτικά, τα διατυπώνω έτσι με τέτοιο τρόπο. Ε, τελικά αυτό ήταν το αποτέλεσμα όμως. Και με αυτή τη συμβαστική τροπολογία ήδη από τώρα έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις τριμερείς με Συμβούλιο και Επιτροπή. Δηλαδή ουσιαστικά εμείς μπορούμε ήδη να αποφασίσουμε ορισμένα, αλλά έχει αρχίσει μια διαδικασία αλλά δεν είναι η άποψη της πλειοψηφίας της Επιτροπής Μεταφορών. Εγώ προσπαθώ πραγματικά πιεστικά τις δύο αυτές θέσεις να τις ε, φέρω πιο κοντά να τη συνδυάσω και να μας εγγυηθείτε ότι στην κατανομή των πόρων θα λάβετε τα μελήματα της Επιτροπής μας υπόψη. Και εμείς να κάνουμε την υποχώρηση για να σου πούμε ότι θέλουμε τις διαδικασίες ανταγωνισμού και στο τμήμα της συνοχής. Γι' αυτό τον καιρό προσπαθούμε με όλους τους ενδιαφερομένους να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό και για τα διαδικαστικά ζητήματα δεν λέω ότι υπάρχουν τώρα ήδη λιμένες αποφάσεις στον τριμερή διάλογο. Λαμβάνουμε υπόψη και αυτά που λέγουν οι δύο ε, συναρμόδιες επιτροπές, αλλά ε, να λάβετε παρακαλώ υπόψη και την Περιφερειακή Επιτροπή. Εμείς έχουμε μια γνωμοδότηση, οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατηθούν μέχρι αύριο και στη δική μας γνωμοδότηση λοιπόν θέλουμε να ε, καταλήξουμε σε συμβιβασμό, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον, ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα. Απλώς θα ήθελα να σας επισημάνω ότι αυτή είναι η σκοπιά και το πρίσμα της Επιτροπής μας. Ο κύριος Σάγκα από την Επιτροπή των Περιφερειών, τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Είμαι Σλοβαίνος. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και για το ότι μου δίνετε το λόγο για να παρουσιάσω την άποψή μου με βάση τη γνωμοδότηση που υιοθετήσαμε στην Επιτροπή μας για το ΔΣΕ. σύγμα ε. ε. Τον Ιούλιο την υιοθετήσαμε την γνωμοδότησή μας με πλειοψηφία. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές υποστηρίζουν αυτό το νέο μέσο. Τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Ε, πώς προετοιμάσαμε αυτή την έκθεση. Ήταν περίπλοκο ζήτημα, κάναμε πολλές διαβουλεύσεις με εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης MOVE. Κάναμε πολλές συνεδριάσεις και με διάφορους ενδιαφερόμενους, με εκπροσώπους τοπικών αρχών και φορέων, επαγγελματικούς φορείς και κλάδους. Είχαμε πολλές επαφές με εκπροσώπους και του Ευρωκοινοβουλίου, με ευρωβουλευτές δηλαδή. Είχα επαφές σε πολλά επίπεδα. Τι λέει η γνωμοδότησή μας. Τρία βασικά πράγματα. Οι επενδύσεις στον, στην ενέργεια, την ψηφιοποίηση και σε όλους αυτούς τους τομείς είναι πολύ σημαντική, ειδικά σε, περίπτωση, σε περίοδους κρίσης. Ε, μας αρέσει ε, η μόχλευση που υπάρχει και θα υπάρξει και ένας πολλαπλασιαστικός παράγοντας, χάρη στον τρόπο χρηματοδότησης. Επίσης, μας αρέσουν και οι προτάσεις για τα ευρωομόλογα. Υπάρχει μεγάλη υποστήριξη για αυτό το μέσο από την Επιτροπή μας. Θα θέλαμε να κάνουμε λοιπόν και κάποιες προτάσεις. Θα θέλαμε να πούμε ότι η εφαρμογή της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος ε, της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής όταν ε, ετοιμάζουμε το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης και όταν ε, επιλέξουμε τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Θα θέλαμε η Επιτροπή να μας εξηγήσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Συνοχής ότι λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές ποσοστώσεις των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Συνοχής και θα πρέπει να σεβόμαστε και τα κριτήρια του Ταμείου Συνοχής. Νομίζω αυτό λέει και το Συμβούλιο και η Επιτροπή Ρέτζιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Περιφερειακή Επιτροπή. Πρέπει να βρούμε ένα συμβιβασμό εδώ, μια συνενετική προσέγγιση που αναγκαστικά είναι συμβιβασμός και ελπίζουμε όλα τα μέλη των συναρμόδιων επιτροπών να συμφωνούν με αυτή την άποψη. Οι δημοσιονομικέ πτυχέ είναι πάρα πολύ σημαντικέ για τι περιφερειακέ και τοπικέ αρχέ. Πιστεύουμε ότι αυτό το μέσο, αυτή η διευκόλυνση θα έχει μεγάλη επίπτωση στου ε, τοπικού προπολογισμού. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ έχουν και νομικέ ευθύνε σε πολλού τομεί. Για αυτού του λόγου θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στη διαδικασία λήψη των αποφάσεων που αφορούν το μέσο αυτό, το ΔΣΕ. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι αυτά τα προγράμματα δεν μπορεί να εφαρμοστούν σωστά εάν δεν συμπεριλάβουμε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην ε, φάση της εφαρμογής. Θα ήθελα λοιπόν να, δώσω, να παροτρύνω τα κρατη να λάβουν υπόψη τους ε, τι διοικητική υποστήριξη μπορούν να προσφέρουν τι υποστήριξη διαθέτουν. Επίσης, σε ό,τι αφορά την αρχή, ε, ο πρώτος που θα ζητήσει θα πάρει και όποιος δεν χρησιμοποιεί κάτι, όποιος δεν προωθεί τα προγράμματά του, ακυρώνται αυτά τα προγράμματα, φοβάμαι ότι αυτό θα είναι μεγαλύτερο εμπόδιο παρά καλό. Αυτά και σε ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε. Πολύ ωραία. από την Επιτροπή Μεταφορών, οι σκιώδεις εισηγητές. Θα σας διαβάσω τον κατάλογο, ανάλογα με το πόσο σηκώσετε το χέρι σας. Mr. Cramer, Mr. Gross, Mr. Alcadrawi, Mr. De Grandes, Mrs. Tico, Mr. Danielis, Mr. Ertog, Ertog, Mr. Kumutsatsos, and from ITRA I have got Mr. Vida Odi. Odi. Θέλετε όλοι να μιλήσετε ή ποιος άλλος θέλει να μιλήσει. Σκιώδης της Ήτρε, εσείς, ναι. Σας καταγράφω. Τους γράφουμε όλους αυτούς. Mr. Prillo's next anyway because Shadow. Yeah. Uh, and... Είναι ο επόμενος, είναι σκιώδης της Ήτρε. Πολύ ωραία. Well, the first is Mr. because a shadow from and... πρώτος, είσαστε σκιώδης εισηγητής της Ήτρε. Σας αφήνουμε να ξεκινήσετε γιατί είμαστε ευγενεί. Τρία λεφτά ο καθένας. Ευχαριστώ μεταξύ, Έχει ξεκινήσει ο, ο μιλητής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο από την αρχή, πρώτος πρώτος. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους τρεις εισηγητές για την έκθεσή τους που βελτιώνει σημαντικά το κείμενο της Κομισιόν και ξεκαθαρίζει ακόμη περισσότερο την πρόταση, ξεκαθαρίζει δηλαδή και τα κριτήρια για να χρησιμοποιηθούν τα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και τα ποσοστά χρηματοδότησης. Η βασική ιδέα που ε, παρουσιάζει το σχέδιο έκθεσης ε, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Δηλαδή, ο σκοπός του μηχανισμού αυτού διευκόλυνση για τη σύνδεση της Ευρώπης θα πρέπει να κινητοποιήσει κονδύλια για προγράμματα τα οποία μπορούν να έχουν μια προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να συγκεντρωθούν οι πόροι για την υλοποίηση προγραμμάτων ε, βάζοντας το ελάχιστο, το μέγιστο κατόφλι στο 1,5%. Έχουμε για πρώτη φορά μια κοινή πλατφόρμα επενδύσεων για τις υποδομές αυτών των τριών βασικών τομέων για την οικονομική ανάπτυξη Ευρώπης. Μεταφορές, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες. Έχουμε αυτό το διατομιακό χαρακτήρα του μηχανισμού αυτού του ΔΣΕ. Ακριβώς γι' αυτό ε, είναι πολύ σημαντικό στο άρθρο 10 να ξεκαθαρίσουμε τη δυνατότητα αύξηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης για τα ε, προγράμματα που έχουν που παρουσιάζουν συνέργειες. Επίσης θα πρέπει ε, να προωθούνται και οι στόχοι του πακέτου κλίματος για τον ορίζοντα Ευρώπη 2020. Θα πρέπει επίσης ε, να ξεπεράσουμε το 10% ε, το ποσοστό χρηματοδότησης όταν έχουμε προγράμματα τα οποία έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Όταν είναι καινοτόμα τα προγράμματα, όταν είναι βιώσιμα περιβαλλοντικά τα προγράμματα Επίσης, θα πρέπει να εντοπίζουμε αυτά τα προγράμματα που έχουν αυτή την ε, ιδιότητα της συνέργειας. Για το άρθρο 7 για την επιλεξιμότητα και τις ε, προϋποθέσεις για την οικονομική βοήθεια, το, η τροπολογία 54 συνάδει απόλυτα με τα όσα λέει ο κανονισμός για τις κατευθυντήρες γραμμές για τις ε, ενεργειακές υποδομές. Ε, για το σημείο Β όμως, ε, πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά τα προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος. Πρέπει να δούμε λοιπόν επίσης και ποια είναι τα προγράμματα που είναι εμπορικά βιώσιμα, αλλά που παρόλα αυτά έχουν ε, κάποιο εμπορικό κίνδυνο για τον ε, επενδυτή. Έχουν δηλαδή μία βαθμολογία κάτω του ελάχιστου για να πάρουν τη συγχρηματοδότηση. Μπορεί να δημιουργηθούν εδώ προβλήματα τη στιγμή επιλογής των προγραμμάτων στον τομέα της ενέργειας που μπορούν να λάβουν τη συγχρηματοδότηση. Σε ό,τι αφορά τι μεταφορές, ε, νομίζω ότι είναι σημαντική η εισαγωγή κάποιων οριζόντιων προτεραιοτήτων για του θαλάσσιου αυτοκινητοδρομού. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ την ολοκλήρωση και τις, των ε, λιμενικών υπηρεσιών και την, ε, να δούμε τι υπηρεσίες παρέχουμε, παρέχουμε στους λιμένες και πώς συνδέονται όλα αυτά με τους θαλάσσιους ε, αυτοκινητοδρόμους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεμπάκερ για τρία λεπτά και παρακαλώ τη γραμματεία να βάλει μπρος το ρολόι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους εισηγητές. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε μια πάρα πολύ δύσκολη έκθεση. Και έχουμε και πολύ δύσκολο δρόμο μπροστά μας και μακρύ. Καταρχάς θέλω να πω ότι Απομένει να δούμε πόσα χρήματα θα διατηθούν για όλη την ευκόλυνση, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε σαν να υπάρχουν τα χρήματα, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Σε ό,τι αφορά τώρα το τμήμα των μεταφορών της όλης υπόθεσης, θεωρώ ότι έχει σημασία εκεί να συνεχίζουμε να πιέζουμε για ίσους κανόνες παιχνιδιού. Ε, ε, αν αρχίσουν τώρα τα διάφορα μέσα μεταφοράς να διαγωνίζονται για το ποιος χρειάζεται περισσότερα κονδύλια και περισσότερη αύξηση, όχι, θα πρέπει με τον ίδιο τρόπο να τους αντιμετωπίσουμε. Ας πούμε, αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι, τα είπαν οι συνεισηγητές ε, και έχουν κάνει ενδιαφέρουσε προτάσεις για ε, τους διαδρόμους. Δεν θέλω να προσθέσουμε τώρα στοιχεία περιφερειακά, τοπικά. Την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Έκλεισε. Συμφωνώ με την τροπολογία 49. Ε, φαίνεται να το συνδέει με τα διευρωπαϊκά δίκτυα ε, μεταφορών, αλλά να το ξανακοιτάξουμε αυτό για τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τι γίνεται και στον προπολογισμό. Είναι πολύ σημαντικό για τη διευκόλυνση που έχουμε αυτό το μέσο ε, και θα πρέπει να λειτουργήσει ε, σωστά. Ε, η 64 τροπολογία βελτίωση τη προσβασιμότητας των υποδομών για τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Συμφωνώ με την πρωτοβουλία, αλλά δεν είμαι ότι είναι του παρόντο 75. Use it or lose it. Αξιοποιήστε το ή χάστε το. Εμ δεν ξέρω, είναι πιο χαλαρή η πρόταση σε σχέση με αυτά που λένε οι συγητέ. Το θέμα είναι να εφαρμόζονται τα προγράμματα στο χρονικό πλαίσιο. Οι θαλάσσιε λεωφόροι είναι επίση ένα σημαντικό σχέδιο και θα πρέπει ε, οριζόντια προτεραιότητα να τη θεωρήσουν οι συγητέ. Είναι καλή βελτίωση. Ε, άλλα σημαντικά θέματα. Ε, καινοτομία, νέε τεχνολογίε μεταφορέ. Χρειάζεται ιδιαίτερη εστίαση και προσοχή και θα πρέπει να το συνδέσουμε και με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα όπω το Horizon 2020. Κατανοώ ότι δεν μπορούμε να προσθέσουμε οτιδήποτε θα θέλαμε να χρηματοδοτηθεί από τη διευκόλυνση και το τελευταίο είναι το πιο λεπτό πολιτικά είναι τα 10 ε, δισεκατομμύρια από το Ταμείο Συνοχής και θα πρότεινα εδώ να παραμείνουμε όσο γίνεται ε, εγκύτερα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εάν ε, αρνηθούμε τα 10 δισεκατομμύρια, δεν θα επιστρέψουν ε, αυτά τα χρήματα απαραίτητο στο Ταμείο Συνοχής, μάλλον θα χαθούν από τον κοινοτικό προπολογισμό, είναι το πιο πιθανό και δεν θα πρέπει. Ξέρω, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης υπάρχουν προβλήματα, αλλά κοιτάξτε τι λέει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, ε, πώς χρησιμοποιήθηκαν τα κονδύλια της συνοχής στις λιμενικές υπηρεσίες και στην πολιτική. Τρία λεπτά. Κύριε Σοντή, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα με τη σειρά μου να συγχαρώ ε, που συνεργάστηκαν ε, πάρα πολύ καλά μεταξύ τους. Διερωτώ με μήπως ε, ξεχνάμε ένα μεγάλο σχέδιο επενδύσεων σε σχέση με τους δημοσιονομικούς ε, περιορισμούς. Υπάρχει τροπολογία 42 που χρειάζεται, ότι, ε, λέει ότι χρειάζεται ένα 3 ε, ευρώ. Ε, ποια είναι η σχέση ανάμεσα στο 1-3 ευρώ και τα 50 δισεκατομμύρια που τελικά δίνουμε ε, μέσω των εκτιμήσεων της Κομισιόν. Αυτά προβλέπει η Κομισιόν. 50 δις. Τελικά κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να εξασφαλίσουμε καινοτόμε χρηματοδοτήσει. Υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη, ειδικά το δικό μου, α πούμε, όπου τον 20ο αιώνα χρηματοδότησαν όλη την ηλεκτροδότηση ας με της υπαίθρου με μία μορφή υποχρεωτικού τέλους. Ξέρω πολύ καλά ότι οι φόροι δεν είναι πολύ έτσι, της μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για τέτοια αν χρειαστεί να επιλέξουμε ανάμεσα στην επιδα... Ε, επιχορήγηση ή σε αυτό το τέλος, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε να υπάρχει αυτοχρηματοδότηση αυτών των δικτύων. Ε, συγχαίρω τους εισηγητές και διερωτώ με αν το κοινοβούλιο μας δεν θα πρέπει να δείξει περισσότερη τόλμη, ειδικά σε αυτό το μεγάλο σχέδιο επενδύσεων ε, του 1-3, που είναι και το αντικείμενο της τροπολογίας 42. Ευχαριστώ πολύ και εγώ τους ηγητές για την έκθεσή τους. Θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω αυτό που είπε ο κύριος Ρικέ. Διασυνοριακή κυκλοφορία, ε, ενίσχυση της ανάπτυξης, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, προγράμματα πιο γρήγορα αυτοχρηματοδοτούμενα. Όλα αυτά είναι ωραία, αλλά τι μας δείχνει εμπειρία. Κανένα από αυτού του στόχου δεν τον έχουμε πετύχει, παρόλο που 30 χρόνια το επιδιώκουμε. Κουρελού είναι η Ευρώπη στο σιδηροδρομικό δίκτυο και πού είναι οι τρύπε τη Γκουρελού στα σύνορα. Και πού είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία πουθενά. Να παραμείνει λέτε το παράρτημα. Ε, θα έχουμε τους παλιούς διαδρόμους. Και μάλιστα εκεί που είναι πιο ακριβό, δεν ε, ε, γράφεται ως διάδρομος, αλλά ο διάδρομος ε, Στοκχόλμη-Παλέρμο πρέπει να περάσει τις Άλπεις, τον Μπρένερ, παρόλο που η Αυστρία τρία χρόνια μπλοκάρει τα έργα γιατί δεν έχει λεφτά. Δεν βγάζουμε τα συμπεράσματά μας, δηλαδή ποντάρουμε σε έργα που ε, κρατάνε χρόνια και δεν ε, δημιουργούν θέσεις απασχόλησης γιατί ε, για να κάνω σύραγγα στις Άλπεις βάζω ένα μετροπόντικα ας πούμε εκεί και δεν δημιουργώ θέσει απασχόλησης. Ε, αν εξηγιάνουμε ε, τους υφισταμένους άξονες και τους αυτοκινητοδρόμους, εκεί θα εργαστούν άνθρωποι. Παράδειγμα, διάδρομος βγαίνει... Ε, ε, Αδριατική από την Πανωνία, το βαθύ, ε, την κοιλάδα εκεί, ε, δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης. Όχι, φτιάχνουν σύραγγα στο Σέμερινγκ, τρυπάνε καινούριο τούνελ και δεν ξέρει κανείς πότε θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Και εκεί μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Ας πούμε το τροχαίο υλικό κάνει θόρυβο, δεν μπορούμε εκεί να καταπολεμήσουμε. Δέκα δισεκατομμύρια λένε για τις ε, υποδομές για να μειωθεί ο θόρυβος από όλο το τροχαίο υλικό στην Ευρώπη φτάνουν 3 με 4 δισεκατομμύρια. Και αυτό αποκλείεται. Στα διευρωπαϊκά δίκτυα παίζει ρόλο ο θόρυβος και αλλού, παντού. Ε, εδώ γιατί δεν το αναγνωρίζουμε και δεν ασχολούμαστε. Γιατί ο διάδρομος στο Χόλμη Παλέρμο δεν περνάει από το Ροστόκ. Γιατί ε, οι δύο σύραγγε τη Ελβετία που ολοκληρώνονται, η μία είναι έτοιμη και άλλη σε δύο χρόνια δεν χρησιμοποιούνται ω εναλλακτική λύση εσκεμένα έχουν επιλέξει διαδρόμους ακριβώς τα προγράμματα και τα έργα των δισεκατομμυρίων. Αυτό είναι υπέρ του κατασκευαστικού λόμπι και υπέρ των τραπεζών, αλλά από πλευρά κοινωνιών ε, ε, η ε, ωφέλεια θα έρθει σε 20 και 30 χρόνια. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα λεφτά. Άλλη προοπτική θέλουμε και πολιτική. Τα 10 τώρα έργα που δεν τα καταφέραμε 30 χρόνια, τώρα σε τέτοιους καιρούς λιτότητας θα τα πετύχουμε. Θα πρέπει να εξαγάγουμε τα συμπεράσματά μας από το παρελθόν, αλλιώς μέλλον δεν θα έχουμε. Αυτή ήταν η Σκιώδης. Τώρα κυρίες και κύριοι, υπόλοιποι βουλευτές. Πόσους έχω? Δέκα ομιλητές. Δύο λεπτά έκαστος, γιατί έχω και τρεις από την Επιτροπή που πρέπει να χωρέσω ε, και ο κύριος Γκρός. Ξέρω ότι θα δώσετε στο καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους εισηγητές. Δεν θα πω στη διευκόλυση στην ουσία. Στην Επιτροπή μας έχουμε σαφή άποψη και για τα έργα μπορούμε να συζητάμε με τις ώρες. Νομίζω ότι μια νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμφωνούμε, αλλά ξέρουμε ότι είναι μεγάλη και η πρόκληση. Τα ίδια τα έργα από τη μια. Μπορούμε να βελτιώσουμε τον κατάλογο, να τον αλλάξουμε, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα έργα αυτά γίνονται σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Επελέγησαν δηλαδή σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να το τονίσουμε. Μπορεί να συζητήσει κανείς προτεραιότητες με τα κράτη-μέλη, αλλά ήταν σημαντική για μένα αυτή η συνεργασία. Γιατί? Γιατί εάν αύριο μειωθούν οι πόροι, Το θέμα δεν είναι να τους εξηγήσουμε πού θα βρουν τα λεφτά, ότι αν περικόψουν θα πρέπει να περικόψουν και έργα, όχι μόνο τα χρήματα. Αυτό είναι το σημαντικό και το λέμε ανέκαθεν και να το πούμε περισσότερο προς τα έξω αυτό. Και βέβαια είμαστε τμήμα ε, των οικονομικών εξελίξεων και του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και βέβαια είναι ε, δύσκολη η οικονομική κατάσταση, αλλά όπως είπε και ο Ντομινίκ Ρικέ είναι πολλές οι προκλήσει και χρειάζονται απαντήσεις πολύ διαφορετικές από άλλα. Ένα τελευταίο που αφορά και συζητήθηκε ιδιαίτερα στην Περιφερειακή Επιτροπή. Εδώ στις μεταφορές θα πρέπει να ξέρουμε ότι μας συμφέρει να είμαστε πάρα πολύ συμπαγείς ε, στην προσέγγιση μας και οι τρεις επιτροπές. Και αυτό αφορά τα 10 δισεκατομμύρια του Ταμείου Συνοχής. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα συμβιβασμού και πρέπει να υπάρχει. Είναι η μέθοδος ΣΕΦ, η κεντρική, ε, αλλά να πούμε και στις χώρες ότι αυτά τα χρήματα που δώσαν εκεί, αν προετοιμαστούν σωστά, θα ε, πιάσουν και τόπο και θα έχουν και απόδοση. Αλλά για να μην έχουμε φαινόμενα του παρελθόντος, ορισμένες χώρες ε, εξασφαλίζουν κονδύλια και δεν τα απορροφούν ποτέ. Θα πρέπει λοιπόν να ε, βρεθεί ένα συμβιβασμό και είναι η μοναδική ευκαιρία που έχουμε απέναντι στο Συμβούλιο παραμείνουμε αξιόπιστοι και να μην χάσουμε ποσοστά που σημαίνουν δισεκατομμύρια. Ευχαριστώ. Μέχρι τώρα δεν έχει τηρήσει κανείς το χρόνο. Όλεθρος. Τρία λεπτά εσύ, Ρόμπερτ, είσαι σκιώδης. Να ευχαριστήσω τους εισηγητές μας ο για τις προτάσεις τους για το δούσου ε. Άκουσα φόβους ότι θα υπάρξει μείωση με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο όλος ο κόσμος μιλάει για περισσότερη Ευρώπη ε, και πιο ομοσπονδιακή Ευρώπη. Αλλά ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός της Ευρώπης μειώνεται από ό,τι φαίνεται. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τους διαδρόμους. Αν χάσουμε τους διαδρόμους αυτούς, όπως λένε οι συγητές, θα χάσουμε την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία αυτό το συζητάμε μονίμως στην Επιτροπή Μεταφορών. Δεύτερον, συμφωνώ με τα σχόλια του κ. Γκρός για τα όσα είπε σχετικά με το Ταμείο Συνοχής. Χρειαζόμαστε ένα καλό συμβιβασμό. Μιλάμε για 10 δισεκατομμύρια ευρώ για τη διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη. Θα πρέπει όμως τα προγράμματα να ολοκληρωθούν από την άλλη. Γιατί θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα. Με βάση την νομοδότηση της Επιτροπής Ρέτζιο, ε, υπάρχει περίπτωση τα 10, τα δισεκατομμύρια ευρώ να ζητήσουν ε, τα κρατημένα να τα επανεθνικοποιήσουν, να τα βάλουν στους προπολογισμού τους. Θυμάμαι μια ιστορία που είπε ο Τζακ Λόντον Έγινε μια μονομαχία. Φανταστείτε να επιστρέψουν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ στα κράτη-μέλη. Τα λεφτά δεν θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε πολλά προγράμματα. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τα 10 δισεκατομμύρια αν θέλετε να προχωρήσει η διευκόλυνση αυτή συνδέοντας στην Ευρώπη. Ο Σαΐτ ε, Αλκαντράου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ηγητές. Το ξέρω ότι υπάρχει θέμα προπολογισμού και είναι μεγάλη ευθύνη του Συμβουλίου. Θα ήθελα κι εγώ να πω ότι είναι πολύ σημαντική η συζήτηση για τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Συνοχής. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να κάνουμε προσπάθειες έτσι ώστε να συμφιλιώσουμε δύο δύσκολα πράγματα. Το ένα, να διαφυλάξουμε ε, τη χρηματοδότηση των χωρών συνοχής από τη μια και από την άλλη, όμως να προσπαθήσουμε να ε, διατηρήσουμε μια κεντρική διαχείριση ε, της Ευρώπης, να μην δώσουμε μια επιταγή ελευκό για τα έργα αυτά. Ε, νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα συμβιβασμού αν κάνει ο καθένας προσπάθειες και επιδείξει καλή θέληση. Και εμείς ε, από την Επιτροπή μας θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ε, στο άρθρο 10 και 17 γίνεται λόγος για συνέργεια μεταξύ έργων τηλεπικοινωνιών και ε, μεταφορών, 10% επιπλέον χρηματοδότηση βλέπετε και καλό είναι αυτό και θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η καλύτερη ιδεώδη κλίδα κατανομής για να μπορέσουν όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης και καλή συνάφεια μεταξύ της διευκόλυνσης ε, αφενός ε, και των κατευθυντήριων γραμμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ας πούμε τι είναι ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ορισμός δηλαδή γιατί έχει διαφορές από έκθεση σε έκθεση και επίσης ε, στους σιδηροδρόμους το θέμα του θρύβου και τέλος να πω ότι για τη συγχρηματοδότηση, συνυπευθυνότητα θεωρώ πάρα πολύ θετικό και τη διαλειτουργικότητα ε, στα τρένα και έργα ε, που προάγουν την κινητικότητα ανθρώπων με περιορισμένη κινητικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βιντάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε ο κύριος Βιντάλ Κουαδράς. Το πρόβλημα χρηματοδότησης μεγάλων έργων στην Ευρώπη δεν είναι καινούριο, αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες έχει επιδεινωθεί κατά πολύ. Υπάρχουν κυβερνήσεις που μείωσαν ε, τις επενδύσεις σε υποδομές με τρόπο δραστικό για να μην πω δραματικό και αυτό είναι εις βάρος και των επιχειρήσεων ε, του κατασκευαστικού τομέα και η τράπεζα είναι σε μια μέγενη που θα πρέπει να δώσει το κάψιμο ας πούμε, για αυτή την υπόθεση. Ε, υπάρχει ένα θέμα αφαιρεγγιότητας και ένα θέμα ρευστότητας στις τράπεζες. Λοιπόν, η έκθεση ζητάει ότι θα, ε, θα πρέπει να βρεθούν καινοτόμε λέει, ε, μορφές χρηματοδότησης θα πρέπει να είμαστε πολύ καινοτόμοι και πολύ εφάνταστοι στην προσέγγιση μας τέτοιους χαλεπούς καιρούς. Και επίσης είναι σημαντικό αυτό που λένε ορισμένες τροπολογίες ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν στρεβλώσεις στην αγορά, τα έργα να φέρουν πραγματική ευρωπαϊκή υπεραξία, να εκμεταλλευτούμε τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων μορφών υποδομών που καλύπτονται από το κανονισμό και υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων μέσων ε, και ε, έργων. Επίσης, όπως λέγουν άλλες τροπολογίες, είναι καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο πρωταγωνιστικό, γιατί είναι και δημοσιονομική αρχή και να ενημερώνεται για τις αποφάσεις που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν εγκριθεί το ετήσιο πρόγραμμα και να γνωρίζει και την ενδιάμεση αναθεώρηση και την εκτοριστέρων αξιολόγηση ε, των αποτελεσμάτων. Τελειώνοντας, Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ δύσκολη καιρή για τόσο φιλόδοξα έργα και ας ελπίσουμε ο κανονισμός αυτός να είναι τμήμα της λύσης. Ευχαριστώ. Η κυρία Φόρτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να μιλήσω γρήγορα και σύντομα. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα σημεία συμφόρηση είναι γνωστό το επιχείρημα ότι πρέπει να ε, το κεντρικό δίκτυο, αλλά υπάρχουν σημεία αυτού του κεντρικού δικτύου που έχουν ε, αποδειχθεί σημεία συμφόρησης σε τεράστιο βαθμό και ίσως να ήταν καλύτερα να επενδύσουμε στο συνολικό δίκτυο ε, ως τρόπο για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα σημεία συμφόρησης. Έτσι λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτά τα σημεία συμφόρησης ε, ε, με επενδύσεις στο γενικότερο δίκτυο. Τώρα, όσον αφορά τα προτινόμενα προγράμματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων και τα λιμάνια. Πιστεύω ότι δεν είναι σημαντικό μόνο το ότι υπάρχει σε ένα λιμάνι, αλλά καθώς επίσης και οι υποδομές που βρίσκονται στο, στην ίδια περιοχή, στην ενδοχώρα. και αυτό που προσπαθούμε σε αυτήν την επιτροπή είναι να ενισχύσουμε το εμπόριο και άρα θα πρέπει να κοιτάξουμε και τα λιμάνια που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για το εμπόριο και βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην περιοριζόμαστε μόνο στα δικά μας. Και τέλος για το ζήτημα της ευρυζωνικότητας που το συζητάμε συχνά στην επιτροπή μου και υποστηρίζω ένθερμα το ψηφιακό θερματολόγιο αλλά πρέπει να ε, είμαστε βέβαιοι ότι υποστηρίζουμε και τις αγροτικές περιοχές, όχι μόνο τις αστικές. Στις αγροτικές περιοχές θα είναι ακόμα πιο δύσκολο και εκεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, ο ιδιωτικό τομέα δεν τις υποστηρίζει επαρκώς. Ίσως λοιπόν εκεί να χρειάζεται η δημόσια χρηματοδότηση ή ίσως με τη μορφή επιχορηγήσεων ή άλλων χρηματοδοτικών μορφών γιατί διαφορετικά θα φτάσουμε σε μια οικονομία δύο ταχυτήτων. Θα έχουμε από τη μια τις αγροτικές περιοχές, από την άλλη τις αστικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και κυρίως στην Κούμπρια θα πρόσθετα εγώ ως περιοχή. Ε, κύριος Δεκράντης για δύο μέτρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μας αρέσει η έκθεση των συγκητών καταρχάς πριτανεύει η αυστηρότητα, η σοβαρότητα και δυστυχώς και ο ρεαλισμός. Γιατί τι να κάνουμε, αυτά έχουμε τώρα. Χρειάζεται έργα υποδομής η Ένωση για να υπάρχει μεγαλύτερη διασύνδεση, ε, ολοκλήρωση της Ένωσης με τις περιφέρειες. Είναι βασική η ιδέα ε, και η ανάπτυξη των δικτύων συνδέεται με αυτό. Συμφωνούμε με τους ηγητές για τη γεωγραφική κατανομή που θα πρέπει να είναι ισορροπημένη. Και τέλος, τα, το Ταμείο συνοχή και η πόρη του ε, βοηθάει στην αύξηση του πλούτου. Θα πρέπει να υπάρξει μια βέλτιστη χρήση των πόρων που έτσι και αλλιώς θα είναι ενιχρή. Γι' αυτό είναι πρόσφορη ιδέα ακριβώ να αναζητήσουμε συνέργειε σε διάφορου τομεί. Υποστηρίζουμε την πρόταση, οι επιδοτήσει κατά προτεραιότητα να πάνε στους διαδρόμους της διασύνδεσης, ε, της διευκόλυνσης συγγνώμη, συνδέοντας στην Ευρώπη. Ε, και Τέλος, θα πρέπει να προωθήσουμε όλες εκείνες τις δράσεις που φιλοδοξούν στη λειτουργικότητα ε, των συνδρομικών ε, μεταφορών. Και τέλος, και τελειώνω Πρόεδρε, ελπίζω να μην κάνει εκπτώσεις στο Συμβούλιο και να είναι αυτά όνειρα θερινής νυχτός. Αν γίνει κάτι τέτοιο, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν θα κερδίσουν αξιοπιστία, αλλά ε, θα χάσουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κορέα Ντεκάμπος για δύο λεπτά. Thank you, Mr. President. I... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν διάβασα προσεκτικά αυτή την έκθεση, δεν είχα το χρόνο, αλλά πιστεύω ότι είναι καλή η δουλειά που έγινε από τους εισηγητές. Η έκθεση αυτή προτείνει για την ενέργεια κάποια πράγματα τα οποία αντιβαίνουν σε όσα εγκρίναμε σήμερα στην έκθεσή μας για την ενέργεια. Σήμερα πήρα την εντολή, μια εντολή μάλλον, ε, για διαπραγματεύσεις. Το Συμβούλιο θέλει να έχει τελειώσει αυτήν την ιστορία μέχρι το Δεκέμβριο. Δεν μπορώ να έχω μια πρόταση που να πηγαίνει προς δύο κατευθύνσεις. Δεν μπορώ να δεχθώ μια τέτοια σχιζοφρονική λύση, όπου οι προτάσεις του άρθρου 15 του κανονισμού μας ε, καταστρέφονται και ακυρώνονται με αυτόν εδώ τον κανονισμό. Είναι αδύνατο να προχωρήσουμε έτσι. Η πρώτη σύσταση λοιπόν που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι να είμαστε συνεπείς. Εγκρίναμε σήμερα ένα νομοθετικό κείμενο. Στην πρώτη ανάγνωση. Δεν μπορούμε να δείξουμε στους εταίρους μας το Συμβούλιο δηλαδή, ότι για θέματα συναπόφασης για το ίδιο θέμα, έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις. Προσοχή λοιπόν, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να ξαναδούμε τις τροπολογίες, κυρίως αυτά αφορούν το άρθρο 54 και το άρθρο 60 που αφορούν την ενέργεια. Προσεκτικοί πρέπει να είμαστε εκεί, γιατί δεν θα έχουμε αξιοπιστεί απέναντι στο Συμβούλιο αν έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις για το ίδιο θέμα. Κυρία Τικάου, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ συγχαίρω τους τρεις εισηγητές. Κάποιες παρατηρήσεις γενικής φύσεως καταρχήν. Είναι σημαντικό να κατανοούμε σωστά τις προσπάθειες, τα προγράμματα δηλαδή, γεωγραφικός πώς προγράμματα για τους διαδρόμους. Για τις νέες χώρες, μην ξεχνάτε ότι αυτές έχουν πιο μεγάλες ανάγκες σε ό,τι αφορά και τους τρεις τομείς, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και μεταφορές. Και όμως ε, είναι πολύ λίγο παρόντα αυτά τα νέα κράτη-μέλη στους ε, διαδρόμους αυτούς. Τώρα, για, τους, ε, για τον τομέα των μεταφορών πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να δούμε ποια λιμάνια και ποιοι θαλάσσιοι διάδρομοι είναι επιλέξιμοι. Σε ό,τι αφορά τα 10 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Συνοχής, πρέπει να προβλέψουμε τους εθνικούς προϋπολογισμούς, ούτως ώστε τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στην πολιτική συνοχή να μην χάσουν αυτά τα κονδύλια. Σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες, τις τηλεπικοινωνίες, το Κοινοβούλιο θα πολεμήσει μέχρι σε σχάτων απέναντι στο Συμβούλιο, ούτω ώστε ο προπολογισμό αυτός να μην μειωθεί δραστικά. Και τέλος, ό,τι αφορά την ενέργεια, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε πιο εμφατικά ότι η τερματική σταθμή υγροποιημένου αερίου είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε αυτόν τον πόρο, ιδίω στη Μεσόγειο, οι χώρε που βρέχονται από τη Μεσόγειο και από τη Μαύρη Θάλασσα. Επίση, να υπάρχει σχέση ανάμεσα στην Κασμία, Κασπία Θάλασσα και στη Μαύρη Θάλασσα. Ο κ. Κουμουτσάκο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε, αυτή η έκθεση είναι εξαιρετικά σημαντική και νομίζω ότι είναι η συνισταμένη όλων όσων συναδέλφων μίλησαν μέχρι τώρα. Θέλω να συγχαρώ του εισηγητέ για την δουλειά που έχουν κάνει, την πολύ καλή δουλειά που έχουν κάνει και να ευχαριστήσω ιδίω του, του δύο ε, εισηγητές τη Επιτροπή Μεταφορών με του οποίου είχα και την τύχη ε, να ε, ανταλλάξω απόψει ω συνεισηγητή στο θέμα των κατευθυντηρίων γραμμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Και υπό αυτή την ιδιότητα χαρακτηρίζω την έκθεση για το Connecting Europe Facility ως οξυγόνο για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Είναι πραγματικά το οξυγόνο για να προχωρήσουν τα δίκτυα σωστά ή λάθος. Και επειδή είναι το οξυγόνο μας ενδιαφέρει και η ποσότητά του και η ποιότητα του οξυγόνου που θα αναπνεύσουμε. Όσον αφορά την ποσότητα, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε μειώσεις που ουσιαστικά θα καταστήσουν την προσπάθειά μας αναποτελεσματική. Την προσπάθεια να διαμορφώσουμε ένα συνεκτικό δίκτυο μεταφορών στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, όσον αφορά την ποιότητα, θα ήθελα δύο μόνο σημεία να θίξω. Ένα αφορά την ανάγκη πιο ουσιαστική στήριξη της ανάπτυξης των θαλασσίων λεωφόρων και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ε, εμείς θα το δούμε και θα το κοιτάξουμε και βεβαίως όσον αφορά τα 10 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Συνοχής προσβλέπουμε σε έναν αποδοτικό, αποτελεσματικό και ρεαλιστικό συμβιβασμό που θα ικανοποιήσει όλες τις πλευρές. Θέλω και πάλι να συγχαρώ τους ηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Mr. Danelis, two minutes, please. Ευχαριστώ κύριος Δανέλης για δύο λεπτά παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους ηγητές για την καλή τους έκθεση. Ε, τρία τηλεγραφικά σχόλια. Πρώτο, θέλω να συμφωνήσω απολύτως με τους συγητές σχετικά με την αναγκαιότητα πρόθεσης των θαλασσίων λεωφόρων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι θαλάσσιες ε, λεωφόροι είναι, ε, συνεισφέρουν εξαιρετικά στην αποσαφήνιση του οδικού δικτύου του ευρωπαϊκού, προσφέρουν οικονομική ανάπτυξη, είναι φιλικές στο περιβάλλον και επίσης για την νησιωτική Ευρώπη αποτελούν μονόδρομο. Δεύτερο, όσον αφορά το ποσό των 10 δις του Ταμείου Συνοχής, Νομίζω ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ αν αποσαφηνίζαμε σε τι συνίσταται η επιπρόσθετη υποστήριξη του σχεδιασμού και της ορίμανσης των έργων που πρέπει να δοθεί στα κράτη-μέλη κατά το σχεδιασμό αυτών των έργων. Τρίτο, σχετικά με τα ποσοστά συγχρηματοδότησης του άρθρου 10, νομίζω ότι όσον αφορά συγκεκριμένα στα ποσοστά για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, εδώ βρίσκει κατάλληλο έδαφος η πρόταση των συναδέλφων Ερτού και Κουμουτσάκου από τη μελέτη, για τη μελέτη κλιματικού αντιχτύπου που προβλέπουν στην έκθεσή τους για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, μόνο που αντί για καθολική προϋπόθεση για όλα τα έργα, αυτή η μελέτη θα μπορούσε να ε, αποτελεί προϋπόθεση για τα έργα που θα λαμβάνουν το επιπρόσθετο 10% ε, χρηματοδότησης ή πιθανόν και για τα έργα μεγάλου προϋπολογισμού. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια και πάλι στους συνεισηγητές. Ευχαριστώ. Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο βεβαίω, ο κύριο Αρτού για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και του ε, δύο εισηγητέ. Ε, Όντω, έχει σημασία και ακούστηκε επανειλημμένα ότι θα πρέπει να έχουμε τα χρήματα διαθέσιμα ε, και θα σας υποστηρίξουμε σε αυτό. Ως συνεισηγητής των κατευθυντηρίων γραμμών θα ήθελα να πω το εξής, ε, που δεν το είδα πουθενά στο έγγραφό σας. Το θέμα των εκπομπών θορύβου και την αντιμετώπιση του θορύβου. Αγαπητοί συνάδελφοι, 80% ε, των εμπορευματικών μεταφορών αφορούν αυτοκινητοδρόμους σε όλη την Ευρώπη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα του θορύβου. Και κάθε ευρώ που επενδύεται στη μείωση των εκπομπών θορύβου είναι σημαντικό επιχείρημα. Ας πούμε, έστω και μείωση 10 δεσιμπέλ σημαίνει μείωση κατά το ίμιση της πρόσληψης, της αντίληψης του θορύβου που έχει ο άνθρωπος. Και το κόστος συγκριτικά είναι μικρό, αγαπητοί συνάδελφοι. Με 1000 ευρώ μπορεί κανείς ε, να επενδύσει ε, σε ένα βαγόνι ε, εμπορευματικό μεταφορών για σιγαστήρα ας πούμε για να μειώσει το θόρυβο στο φρένο. Και τέλος, να δώσω και ένα παράδειγμα. Την Ελβετία 1,1 δις ε, επένδυσαν μόνο οι Ελβετοί για τις εμπορευματικέ μεταφορές και το αποτέλεσμα ήταν μεγαλύτερη ποιότητα ζωής, μικρότερο κόστος στο σύστημα υγείας, καλύτερο περιβάλλον και κυρίως μεγαλύτερη αποδοχή στα μάτια των πολιτών. Γιατί αν δεν είναι δεδομένη αυτή η αποδοχή, τότε δεν χρειάζεται να συζητάμε καν όλα αυτά τα προγράμματα και τα έργα, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να τα επιβάλλουμε. Απλούστατα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Ερτού, η Κομισιόν. Ξέρετε πολύ καλά πώς η αυτοπιθαρχία επέδειξαν οι ευρωβουλευτές, ελπίζω και εσείς. Δύο λεφτά ο καθένας. Ο κύριος Πακέ, ο κύριος Διγκράφ και ο κύριος Βινουά μετά. Ο κύριος Πακέ, δύο λεφτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θαυμάσια έκθεση. Είναι μια καλή πολιτική βάση για να συζητήσουμε και με το Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε μια τέτοια έκθεση Είμαστε ευγνώμονες προς τη δουλειά που κάνατε. Ευγνώμονες και προς τους τρεις σας και εσάς συνάδελφοι, τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές για τις παρεμβάσεις σας. Ε, βελτιώνεται πραγματικά το κείμενο της ε, Κομισιόν. Έχουμε κάποια οριζόντια θέματα, ε, κάποια είναι τεχνικά. Αν συμφωνείτε θα τα πω κατευθείαν στους εισηγητές και στη γραμματεία, όχι εδώ. Θέλω να σημειώσω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για τη δουλειά που έγινε για τις συνέργειες. Ε, γιατί αυτό είναι μία από τις βασικές, ε, τα βασικά σημεία, τη βασική λογική της διευκόλυνσης αυτής. Το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστούν. Ε, για τα διάφορα σημεία της επιτροπολογίας τώρα, προφανώς εδώ είμαστε στην παραδοσιακή συζήτηση για το πώς θα εφαρμόσουμε τα μέσα της επιτροπολογίας και νομίζω ότι φαντάζεστε ποια θα είναι η θέση της Κομισιόν. Είναι η παραδοσιακή, δεν χρειάζεται να επανέλθω. Η αναφορά στην εκτελεστική υπηρεσία του, του TNT, του οργανισμού αυτού, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα για, την, για τις μεταφορές. Είναι σημαντικό να λειτουργήσει αυτή η υπηρεσία, ούτω ώστε οι Βρυξέλλες να υποστηρίξουν τα κράτη-μέλη για να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των μέσων αυτών για τις μεταφορές το κείμενο το δικό σας βελτιώνει το δικό μας. Υπάρχουν πολλές καλές ε, τροπολογίες, άτομα με ειδικές ανάγκες, θαλάσσες, ε, λεωφόροι κτλ. Για το θόρυβο και την καινοτομία ένα σχόλιο. Είναι πολύ σημαντική τομή στην πρόταση της Κομισιόν. Είμαι διχασμένος γιατί από τη μία χαίρομαι που εστιάζεται πολύ στην υψηλότερη δυνατή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, όπως λέει το παράρτημα 1, αλλά υπάρχουν και κάποια υπιότερα μέτρα και που θα έχουν πολύ σημαντική επίπτωση. Σημαντικό και αυτό. Φυσικά υπάρχουν και κάποια τεχνικά μέτρα για τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα και τις επιχορηγήσεις και το πώς αλληλεπιδρούν τα μέσα στα δε. Θα τα δούμε αυτά διμερώς. Δέκα δευτερόλεπτα, Πρόεδρε, για αυτό που είπε ο κύριος Πίπερ και το επανέλαβαν πολλοί ευρωβουλευτέ για τα δεκαδεί και τη σχέση αυτών των δεκαδεί με τα διάφορα μέσα πολιτικών. Οι αρχέ που ανέφερε ο κ. Πίπερ, ο κ. Γκρό και άλλοι. Πιστεύουμε ότι, εμείς, ότι η πρόταση για τη διευκόλυνση λαμβάνει υπόψη όλε αυτέ τι προτάσει. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να το πετύχουμε αυτό, αλλά αν μπορούν οι δύο επιτροπέ να βρουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να προχωρήσουμε, θα ήμουν ευγνώμων. Σοκαριστικά δύο λεφτά, κύριε Ντιγκράφ. Ε, ελπίζω να είστε καλύτερος χρονικά. Ε, τα 45 δευτερόλεπτα που σα πήρε ο κύριο Πακέ θα προσπαθήσω να στα δώσω μιλώντας λιγότερα για τις ενέργειες. Για το ψηφιακό κομμάτι της διευκόλυνση. Αν θέλετε να έχουμε μεγάλη α, επίπτωση, ε, θα πρέπει να κάνουμε επενδύσεις ε, στις τηλεπικοινωνίες. Είναι σημαντικό αυτό. Επίσης, ε, αυτό που λέει η εκθεσή σας για τη διαλειτουργικότητα, για την τεχνολογική ουδετερότητα, για το άνοιγμα των δικτύων, για την προστασία της ε, πολιτικής κοινωνίας Ευρώπης, ε, ο Επιτροπός μου ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτές τις αρχές. Θέλουν να εφαρμοστούν και το τελευταίο σημείο, κύριε Πρόεδρε, για την σημασία των χρηματοδοτικών μέσων. Συμμεριζόμαστε την άποψη των εισηγητών ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε ε, με χρηματοδοτικά μέσα την ε, ευρυζωνικότητα ε, δεδομένου του στοιχείου της μόχλευσης και θα πρέπει ακριβώς για να προχωρήσει η χρηματοδότηση να υπάρξει και ιδιωτική επένδυση, ιδιωτική χρηματοδότηση. Ένα ευρώ θα δώσουν 5 με 10 ευρώ επενδύσεις τελικά χάρη στο στοιχείο της μόχλευσης. κύριος Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σε τρία σημεία θα περιοριστώ. Πρώτο, τροπολογία 47 όπου αναφέρεται ότι 80% ε, θα πρέπει να πηγαίνει στα χρηματοδοτικά μέσα ε, της ενέργειας, το 80% του προπολογισμού της ενέργειας. Ε, δεν είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο. Έχουμε προβλήματα και χρειαζόμαστε περισσότερες ε, ε, δαπάνες για να διασυνδέσουμε την Ευρώπη με δίκτυα παντού ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και ολοκλήρωση της αγοράς. Το 80% όμως δεν είναι κάτι το οποίο εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και θέλουμε το αντίστροφο, 80% ε, ε, ενίσχυση και 20% από το χρηματοδοτικό μέσο. Η ε, τροπολογία 54, είδαμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής ΙΤΡΕ, μηχανισμός το πρωί και την υποστηρίζουμε, άρα δεν χρειάζεται να έχουμε επικαλύψεις και η τροπολογία 54 ε, νομίζω μάλλον πρέπει να ξεχαστεί. 67-68 τροπολογίες για την ένταση βοήθειας για τη χρηματοδότηση. Εδώ μπορεί να υπάρχουν μεγάλα προβλήματα για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, διότι εκεί είχαν συνηθίσει να έχουν ενίσχυση από τα διορθωτικά ταμεία ε, με υψηλή ένταση και πάλι πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να διασυνδεθεί αυτή η περιφέρεια της Ευρώπης, ειδικά στο φυσικό αέριο, κατανοείται όλοι τι εννοώ και είναι απολύτως ε, απαραίτητο να σταματήσουν οι ενεργειακές νησίδες που υπάρχουν εκεί και η επένδυση είναι ακόμα ε, χειρότερη. Γιατί ε, εάν γίνει καλύτερη διασύνδεση θα πέσει η τιμή της ενέργειας. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό θέλουμε μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες υποδομές. Ευχαριστώ. Οι εισηγητές μας. Ένα λεπτάκι ο καθένας. Θέλετε οπωσδήποτε να μιλήσετε. Η κυρία Βαλεάν πρώτη. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι για τα καλά σας λόγια. Ανείχνευσα μια κοινή προσέγγιση ε, για την έκθεση αυτή και χαίρομαι πολύ που όλες οι τροπολογίες και η συνεργασία μας θα είναι ε, επικοδομητική. Για τα τελευταία σχόλια της Επιτροπής να πω ότι δεν με εκπλήσουν. Έχουμε συζητήσει κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της έκθεσης. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα έχω πει στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας ότι Εάν έχει κανείς μόνο 10 δισεκατομμύρια και πρέπει να επενδύσει 200, αυτό δεν λύνεται βάζοντας το 80% των χρημάτων σε ενισχύσεις. Γιατί ενισχύσεις, επιδοτήσεις, ε, ε, επενδύσεις και μετά χάνονται. Δεν υπάρχει υπεραξία. Εδώ δίστανται οι απόψεις μας και οι στρατηγικές μας. Και ε, το υποστηρίζω. Ο κύριος Ρικέ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη βοήθειά τους, για τις παρατηρήσεις, για τη συνεργασία. Ε, θα, τους... θα ξανάρθω σε επαφή μαζί τους ούτως ή άλλως. Ε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Δύο πράγματα που ακούσαμε ξανά και ξανά ήταν ότι ο προπολογισμό αρκεί. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να κάνουμε μια πολιτική μάχη εδώ πέρα, απέναντι στο Συμβούλιο, αλλά και να είμαστε ενωμένοι, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε τον καλύτερο τον προπολογισμό. Δεύτερον, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που υπόθηκαν από τον Πίπερ και από τον Γκρός, ότι θα πρέπει όντως να βρούμε ένα συμβασμό με τη Ρέτζη. Γιατί δεν είναι λογικό να πάμε στον τριμερή διάλογο και ο ένας να λέει τα μεν και ο άλλος τα λέει. Χωρίς να πω σε λεπτομέρειες, νομίζω ότι είμαστε στην καλή κατεύθυνση καλό θα ήταν να βρούμε, και μπορούμε να το κάνουμε, να βρούμε μια θέση που θα ικανοποιήσει και τους δύο, και εμάς και τη Ρέτζη. Όλα τα θα τα συζητήσουμε. Λινές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά όλους τους συναδέλφους που είχαν την καλοσύνη να κάνουν προτάσεις και θα επιλουτίσουν φαντάζομαι με αντίστοιχα με τους, ε, όλες ευπρόσδεκτες. Θέλω να πω ότι σε σχέση με την ανάγκη αυτή να είμαστε ενωμένοι ως Κοινοβούλιο στη συζήτηση απέναντι στο Συμβούλιο, στα δημοσιονομικά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη όλες οι δεσμεύσεις που ισχύουν σήμερα και θα πρέπει δηλαδή να εργαστούμε στην πρώτη εντολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μπορεί να μην μας άρεσε, αλλά τουλάχιστον διέσωσε αυτό το μέσο ε, απέναντι σε κάποιους συναδέλφους που θεωρούσαν ότι καλό θα ήταν να καταργηθεί εντελώς και οριστικά. Συμφωνώ λοιπόν με αυτά που είπατε, αλλά θα πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο για να καταφέρουμε μια γενική ενότητα και των τριών επιτροπών ε, που ασχολούνται με τη δημοσιονομική αυτή πρόταση. Ευχαριστώ. Πριν σας πω τα τυπικά, προθεσμία κατάσταση τοπολογιών, θέλετε να προσθέσετε τίποτα κυρία Πρόεδρε. Όχι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ε, θυμίζω στα μέλη ότι... Η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στις 12 Απριλίου ότι γνωμοδοτήσεις ε, και εκθέσεις δεν θα πρέπει να περιέχουν στοιχεία δημοσιονομικά. Οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνετε τροπολογίες για αύξηση μείωση των ποσών στη διευκόλυνση. Ωστόσο οι επιτροπές θα μπορούσαν να εγκρίνουν τροπολογίες ε, για την σχετική κατανομή, ποσοστά δηλαδή και μερίδια ε, χωρίς ποσά. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών τώρα 4 Οκτωβρίου θα τη συζητήσουμε στις 5 Νοεμβρίου τις τροπολογίες που θα μας δεχτεί η Ήτρε λοιπόν και ε, κοινή ψηφοφορία στις 27 Νοεμβρίου στη ΔΕΟ αν δεν πέσει καμιά άλλη οθόνη, ε, ε, ε, ποστούν ρογμές οι τείχοι, θα πάει τον Ιανουάριο το 2013. Σας ευχαριστώ για την πειθαρχία, για το χρόνο. Είναι σημαντικό αυτό ε, και ευχαριστώ τους συναδέλφους της Ήτρε που ήρθαν εδώ και τους διερμηνείς για τη δουλειά τους. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Λύεται η συνεδρία σας.